Έχετε το λόγο κύριε Σέντερ, είστε ο πρώτος. Λοιπόν, επεξηγήση ψήφου, οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να μα τα πείτε. Για την ε, έκθεση Προβέρα.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 ταραχές στην Τινησία, στην Αίγυπτο και σε πολλές άλλες αραβικές ε, χώρες οδήγησαν σε μαζικά μεταναστευτικά ε, ρεύματα προς την Ευρώπη. Είναι τεράστια πρόκληση αυτή για την Ευρώπη. Θα πρέπει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και ότι χρειάζεται αντιμετώπιση σωστή και κοινή. με αλληλεγγύη θα πρέπει να φροντίσουμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα εξωτερική πίεση αυτή και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκρινε πολιτική για να αποκρουστούν ε, αυτές οι καταστάσεις. Επίσης χαίρομαι για την απόφαση ε, του Κοινοβουλίου να ενισχυθεί ο ρόλος της Frontex. Εμείς οι φιλελεύθεροι το επιδιώκαμε αυτό πάρα πολύ και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Τώρα αυτό που λείπει τι είναι. Οικονομική πόρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Ο κύριος Αρλάκη είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί είναι ένα πρώτο βήμα για μια τέτοιου είδου κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που προκύπτει από την αστάθεια στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικό το Κοινοβούλιο να υψώσει τη φωνή του ε, κατά αυτού του ιστερικού οράματος της πλημμυρίδας μεταναστών που θα καταφτάσουν από τον Νότο. Εμείς δεν θα πνιγούμε από εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τους χώρους τους λόγω πολιτικών προβλημάτων και ταραχών. Πολλοί φοβούνται πως οι ετούντες άσυλο φτάνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς ε, με σκοπό να μάλλον με αποτέλεσμα να καταρακώνουν τα συστήματα μας πρόνοιας. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε την μεταναστευτική πολιτική μας, αλλά τα γεγονότα δεν συνηγορούν πέρα αυτής του καταστροφικού οράματος. Μάλλον που 40% έχει μειωθεί η μετανάστευση ε, τα τελευταία 10 χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Γιακολίνο είναι ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ υποστήριξα και ψήφωσα, ψήφισα ε, το, το έγγραφο του συναδέλφου Προφέρα γιατί πιστεύω ότι αποτελεί ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και μάλιστα προβλέπεται και στο άρθρο 80 και πιστεύουμε ότι δείχνει μια καλή και καθαρή ματιά ε, για, την, ε, για τις χώρες ε, οι οποίες στη Βόρεια Αφρική αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και όσον αφορά τα ανθρώπινα και όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, τις ε, ε, σχέσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και τους οργανισμούς που δρούν επιτόπου, όπως ας πούμε Αραβικός Σύνδεσμος κλπ. Ελπίζουμε ότι τα βήματα προς τα εμπρός θα ληφθούν και μέσω ομοιογενών και ισορροπημένων αποφάσεων που θα βοηθήσουν και την κοινωνία και την οικονομία που θα πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να υπάρξει διαρκής και συνεχής ανάπτυξη. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να δηλώσω ότι λόγω της αστάθειας στην περιοχή αντιμετωπίζουμε μια πραγματική πρόκληση από τις μεταναστευτικές ροές είναι μια πρόκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από άτομα, ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική ιστορία το καθένα και που μετακινούνται για το λόγο αυτό. Στην Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με συμπάθεια και με την ε, βούληση να τους βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει ειρήνη, σταθερότητα στην ε, περιοχή μας. Ε, υπάρχουν δυνατότητες ανέληξης και συστήματα θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής να λυθούν όταν δημιουργούν προβλήματα εσωτερικής πολιτικής. Δεν χρειαζόμαστε μόνο αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και ένα ε, ενεργό πλαίσιο στην Ευρώπη που θα συμπεριλάβουμε την ε, εμπορική, πολιτική, την κλιματική αλλαγή, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ε, εξωτερική πολιτική όλα αυτά, αν συνδυαστούν, θα μας δώσουν τον τρόπο να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές ε, συχνά αναφέρει μα ποια προ πρόβλημα μπορεί να έχει μια χώρα μεγάλη 60 εκατομμυρίων ανθρώπων να υποδεχθεί ορισμένε δεκάδε ή εκατοντάδε ε, μεταναστών. Να απαντήσω ω εξή. Πρώτον, πολλοί από αυτού του μετανάστε θέλουν να φτάσουν σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, τα δύο τελευταία χρόνια έφτασαν ε, λιγότερο από 4.000 άνθρωποι μετά από συμφωνίες με τη Λιβύη και την Τινησία. Τους τελευταίους μήνες μετά τα πρόσφατα γεγονότα έφτασαν 22.000 άτομα. Ε, πρώτον υπάρχει η πίεση των οικονομικών μεταναστών από την ε, Τινησία που δεν μπορεί να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά ε, στην τοποθεσία Βεντιμίλια η Γαλλία επαναπροωθεί τους μετανάστες γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση αυτών των μεταναστευτικών ροών είναι επίγουσα θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε συμφωνίες με, τους χώρες, με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ε, μετανάστες αυτοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σινκλέρ ζητάει διαδικαστικό. Ευχαριστώ πρόεδρε, διαδικαστικό ναι. Εδώ στο ημικύκλιο Πρέπει να συζητούμε και να σεβόμαστε ο ένα τον άλλον. Αλλά όταν έχετε δύο προέδρους πολιτικών ομάδων σε ιδιωτικέ συζητήσεις, όταν ε, οι άλλοι συνάδελφοι μιλούν, τι σεβασμό δείχνει αυτό στους συναδέλφους. Um, Κύριε Ντόλ. Κύριε Λυπάμαι. Μα ζήτησαν να δώσετε εσείς το παράδειγμα. Ο κύριος Ούτζας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα αποσαφηνίζει λίγο την κατάσταση όσον αφορά τι μεταναστευτικέ ροέ και η ενίχυση τη Frontex επίση μπορεί να θεωρηθεί ε, κάτι θετικό κατά την ίδια έννοια και το, η έκβαση τη ψηφοφορία. Όμω πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη διαφάνεια από πλευρά και σαφήνεια από πλευρά των κρατών μερών, γιατί η πρόκληση αφορά βεβαίω <clears throat> τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την πολιτική των κρατών μελών Πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει διαφάνεια στις πράξεις των ε, χωρών έχουμε την πολιτική της Ιταλικής ε, κυβερνήσεως, με, κυβερνήσεως που με πολύ ε, ε, ε, αμφιλεγόμενο τρόπο προσπάθησε να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό κύμα στη Λαμπεντούζα. Αφέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί ε, στην τύχη τους που σε άλλη περίπτωση από άποψη ανθρωπιστική αλλά και νομική θα έπρεπε να είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει και το νομικό ζήτημα να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Μουσκαρντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι πολλές μεταναστευτικές ροές προέρχονται ή οφείλονται ε, από την αστυνομία αστάθεια γιατί έτσι ορίζουμε ε, την, ε, τον, ε, τους, την ανεξελεγκτή βία, τις εξεγέρσεις, τις σφαγές, τους εμφυλίους πολέμους, αυτή τη μιζέρια στην οποία έχουν καταδικαστεί αυτοί οι λαοί με τη σφραγίδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει βεβαίως και η επιθυμία για ελευθερία και για δημοκρατία. Ε, πιστεύω ότι εγκρίναμε σήμερα μια σωστή έκθεση για εργαλεία τα οποία ε, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουμε και την αστάθεια. Αναρωτιέμαι ποια είναι η σωστή εξωτερική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί όταν ε, δεν δείχθη κανένα δείγμα εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το θέμα της νησία ε, κυρίως δε της Λιβύης. Ο καθένας καθένα ή κάθε χώρα κινήθηκε μόνη της και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μία εσχρή εικόνα θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γιατί και η υποδοχή των ε, μεταναστών δεν είναι αυτή που θα οφείλαμε. Ακόμα και τα όσα συμβαίνουν στην Λαμπεντούζα είναι ένα μονάχα δείγμα. Θα πρέπει τελικά να αποκτήσει μια αξιόλογη ευρωπαϊκή πολιτική, άξια του εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, άξια του ονόματος της εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Βανέκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αποχή ψήφισα στην έκθεση Προβέρα. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει σαφήνεια. Προτείνουν τα πάντα, λένε τα πάντα ε, και ε, καμιά φορά κάποια λογικά και είναι αξιοπρόσεκτο αυτό, αλλά τελικά είναι η πλήρης πολιτική ορθότητα πουθενά σε καμία παράγραφο, σε καμία υποπρόταση δεν αναφέρεται στη μετανάστευση, τη νέα μαζική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που είναι υπερβολικός ο πληθυσμός και όλοι θέλουν να πάνε στη Δυτική Ευρώπη. Πουθενά δεν το αμφισβητεί αυτό, δεν τολμάει. Η χώρα μου, η Φλάνδρα, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συντριπτική πλειονότητα των Φλαμαδών δεν θέλουν και νέα μετανάστευση, ιδιαίτερα από χώρε με πολιτισμό και ε, θρησκεία που είναι στο αντίποδα τη δική μα. Κάποια στιγμή θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούει του πραγματικού Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα με βράχη πρόθεσμα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ε, Μεσογείου και ε, να ενισχυθούν ε, εργαλεία όπως η Frontex. Όμως μακροπρόθεσμα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέε θέσει στις χώρες προέλευση των ανθρώπων αυτών ε, και να διαχειριστούμε καλύτερα επομένως μεταναστευτικέ ροέ. Πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να βελτιώσουμε πραγματικά ε, το άνοιγμα των αγορών μας ξεκινώντας από χώρε όπως η Αίγυπτος και η Τινησία. Ήρθε η ώρα επίση να ανοίξουμε διάλογο όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Έχουμε το παράδειγμα της Τουρκίας ε, και την επιτυχία, την επιτυχή έκβαση της Τελωνιακή Ένωσης και τα απαραίτητα μέτρα τα οποία ε, υποβοήθησαν και την, ε, τον εκδημοκρατισμό. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και ειδικών τελωνιακών συμφωνιών με τις χώρες της Μεσογείου. Θα τελειώσω λέγοντας ότι ε, θα πρέπει να καλέσουμε το Συμβούλιο άμεσα να εγκρίνει ε, την ε, συνθήκη για την πανμεσογειακή ρίζα προέλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σοχάναν, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η βασική αρχή αυτή τη έκθεση είναι λανθασμένη. Το ότι η μετανάστευση αποτελεί ε, προϊόν απελπισία και φτώχεια μπορεί βέβαια να θεωρείται πιστικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν αληθεύει. Γιατί ξέρουμε ότι είναι οι προσδοκίες των ανθρώπων που δημιουργούν ε, αυτά τα ρεύματα. Είδαμε τι έγινε στην Τινησία. Ήταν μετά την κατάρρευση της δικτατορίας που ξεκίνησε το μεγάλο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα. Γιατί φεύγει ο κόσμος εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του για την ευκαιρία, κυνηγώντα την ευκαιρία. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε μακρόχρονη διαρθρωτική ανεργία θέλουμε να φέρουμε και άλλους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε Τέσσερα εκατομμύρια ανέργους, οι οποίοι είτε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, είτε μειωμένα επιδόματα απασχόλησης και ξαφνικά ε, βλέπουμε ε, εκατοντάδες ε, και χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται και να παίρνουν θέσεις εργασίας από αυτούς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παγιδευτεί, παγιδευτεί στην ανεργία. Αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να αναθεωρήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε την πολιτική πρόνοια και όχι να ανοίξουμε τις θύρες Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σκαμάλ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται όταν αναφερόμαστε στην ε, μετανάστευση ε, δηλαδή ότι ε, αποφασίζει κάποιος να μετακινηθεί από μία χώρα στην άλλη ε, με μεγάλες δυσκολίες. Αφήνει κανείς ε, τη ζωή του, τους γονείς του, την κοινωνική του ζωή χωρίς να ξέρει αν θα τους ξαναδεί κάποτε. Και παρόλα αυτά προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες οι άνθρωποι αυτοί και πολύ συχνά το κάνουν πάση θυσία γιατί προσπαθούν, προσπαθούν να ξεφύγουν από κυβερνήσεις τις οποίες πλέον δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, και τις κοινέ πολιτικές που έχουμε. Έχουμε ας πούμε πολιτική αλληλείας που επιτρέπει σε μεγάλα αλλιευτικά σκάφη ε, να ψαρέψουν σε άλλα ύδατα αφήνοντας σε απόγνωση τους ντόπιου ψαράδες. Στην Αφρική. Και ε, με τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να αφήσουν τις χώρες τους και να έρθουν εδώ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους και να τους βοηθήσουμε λοιπόν με νέα μέτρα να μείνουν εκεί. Στην έκθεση Γέγκλε, 8 ομιλητές. Ο κύριος Ρόντα, πρώτος και πάλι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να προστατεύουμε όχι μόνο τις γυναίκες αγρότησες αλλά και τους αγρότες, τους άνδρες που εγκαθίστανται στις γεωργικές περιοχές. Χρειαζόμαστε ενισχυμένη γεωργία στην Ευρώπη, ποιοτικά τρόφιμα παντού και για να το εξασφαλίσουμε θα πρέπει να βοηθήσουμε τον κλάδο αυτό που δημιουργεί και θέσει απασχόλησης αλλά και απασχολούνται οικογένειες ολόκληρες στη γεωργία. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να αναπτυχθεί η ύπεθρος, ε, ε, όχι νέες ποσοστώσεις και τεχνητές αποφάσεις που θα επιβάλλουν κάποιες καταστάσεις στη Γεωργία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό που πρέπει να στέλνουμε για τις αγρότησες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριος Πυρίλο. One minute. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στον ε, γεωργικό τομέα και στην Ήπεθρο, οι γυναίκες πάντα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. 42% ε, αντιπροσωπεύουν από την εργασία, 27 εκατομμύρια εργαζόμενες. Ε, παρά αυτό το υψηλό ποσοστό γυναικών, δεν εκπροσωπούνται καλά αυτές στους, στις οργανώσεις του κλάδου και επομένως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν δικαιώματα στι γυναίκε αυτέ, όπω α πούμε η απαραίτητη κοινωνική κάλυψη. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα έτσι ώστε να καλυφθούν ε, αυτέ οι ε, λήψει και να δημιουργηθούν μηχανισμοί όπω αυτοί που έχουν δημιουργηθεί στην Καλαβρία και σε άλλε περιοχέ τη Ιταλία. Θα πρέπει να επίσης ταυτόχρονα να εξεταστεί και το γεγονό τη γενικευμένη εξόδου από την Ήπεθρο προ τι μεγάλε πόλεις, δημιουργία υποδομών, στήριξη των περιοχών, δημιουργία νέων δομών, κατάλληλων και προσαρμοσμένων στη νέα ζωή και στις νέες συνθήκες διαβίωσης. Ευχαριστώ πολύ. Γιάρα. Κύριε Πρόεδρε, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Υπέθρο έχουν αλλάξει ε, λόγω και της δημογραφίας και της αστιφιλίας και των ριζικών αλλαγών. Αν θέλουμε όμως να παραμείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο και οι γυναίκες θα πρέπει να ενισχύουμε ε, τους αγρότες και να λαμβάνουμε πολύ περισσότερο υπόψη την πραγματικότητά τους. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και αυτή τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιες οι γυναίκες μεμονωμένες ή και γυναικείες οργανώσεις ε, διαμόρφωσαν αυτή την αλλαγή και την ε, παρακολούθησαν. Και η συγγήτρια κυρία Γέγλε ακριβώ, τόνισε αυτό το στοιχείο στην έκθεσή της, το έχει διαπραγματευτεί πάρα πολύ σωστά και είναι σημαντικότατη αυτή η έκθεση γιατί αν θέλουμε να απτύξουμε την Ήπεθρο δεν αρκούν κάποιες υποδομές ή κάποια διαμόρφωση της υπαίθρου για τον τουρισμό θα πρέπει να εγκαθίστανται οικογένειες και εκεί χρειάζονται και γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, Mr. Ο κύριος Βοητσικόφσκι. Στηρίζω. Στηρίζω την e, έκθεση της κυρίας Τσίγκλη, γιατί ένας από τους λόγους είναι πως αναφέρεται στους απαραίτητους πόρους που χρειάζεται η Γεωργία. Νομίζω πως η λιτότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εις βάρος της ΚΑΠ. Εάν λοιπόν οι περιοχές της Υπέθρου και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί δεν στηριχθούν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βελτιώσουμε την κατάσταση και των γυναικών και των νέων και θα είναι δύσκολο να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να ζήσουν εκεί. Θα είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε και να πετύχουμε στόχους όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση τροφίμων, η καλή ποιότητα αυτών. Λοιπόν, θα ήθελα να απευθύνω την εξή έκκληση. Τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας να μην λειτουργήσουν εις βάρος της ΚΑΠ. Gracias, presidente. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι θεωρώ ότι συμβάλλει στην καταπαλέμηση της αδιαφάνειας ε, ώστε να δοθεί περισσότερο φως στη συμβολή των γυναικών στην Ήπεθρο. Αλλιώς δεν θα ήταν δυνατό ούτε στο παρελθόν αλλά ούτε και στο μέλλον να διατηρήσουμε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν την κοινωνική συνεισφορά και να αναγνωρίσουμε και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Η καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του φύλου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην κοινή, στη, στην, κοινή γεωργική πολιτική και να ενθαρρύνουμε και την ψηφιοποίηση της Ήπεθρου ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ του άστεως και της υπαίθρου. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη δουλειά των γυναικών και σε επίπεδο παραγωγικό αλλά και σε επίπεδο υποβοθητικό. Πρέπει να αναγνωρίσουν τη συμβουλή των γυναικών στην προστασία των ηλικιωμένων και στη φροντίδα των παιδιών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουσκαρδίνη παρακαλώ. Υπάρχει το 42% των γυναικών ε, και στα 26 εκατομμύρια υπαλλήλων και το 29% των επιχειρήσεων. Ε, πράγματι αυτό ισχύει, άρα δηλαδή η δική μας η παρουσία όμως ε, σε άλλες κατηγορίες είναι σχεδόν μηδενική. Αυτό λοιπόν δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε φυσιολογικό γιατί είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη έκφραση στις γυναίκες κυρίως στο γεωργικό τομέα να βρει τις ε, κατάλληλες λύσεις για να διασφαλίσει την οικονομική δραστηριότητα. Να υπάρχει ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων, προστασία των γυναικών και αναγνώριση του ειδικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στη Γεωργία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προωθήσει την συνεχή του εκπαίδευση. Και ένα θέμα, ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Εμείς συμμεριζόμαστε τις προτάσεις της εισηγήτριας για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά όργανα του γεωργικού τομέα. Θέλουμε να στηρίξουμε ε, πρωτοβουλίες ε, κοινωνικής προστασίας, κυρίως όσον αφορά τη γεωργία οι γυναίκες λοιπόν οφείλουν να την χάνουν αναγνώρισης κυρίως μέσα από την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλιώς η μεταρρύθμιση είναι περιττή και δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα νυφάλιο μέλλον χωρίς να υπάρχει η καινοτομία και η εκπροσώπηση των γυναικών στη γεωργία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την σειρά Life and House της οποίας ο πρώτος ήρωας είχε γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 70. Αισθάνθηκα όπως και εκείνος όταν διάβαζα τον κατάλογο των ψηφοφοριών σήμερα. Βλέπω να προωθούνται, να προωθούνται πολιτικές για τις γυναίκες, ειδικέ χορηγήσεις στην Τσεχία και άλλα θέματα που ομολογώ δεν θα θεωρώ τόσο σημαντικά ως αυτά που θα έπρεπε να απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο στασιπληθωρισμός και ο κίνδυνος χρεοκοπίας ορισμένων χωρών. Φοβάμαι ότι όλα αυτά οφείλονται σε εσφαλμένες πολιτικές. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τις οικονομίες και να επιτυχαίνουν αποτελέσματα με ανακατανομή των πόρων. Τα 27 κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παίρνει χρήματα από τους φορολογούμενους και να τους δίνει σε εκείνους που απειλούνται από χρεοκοπία, διότι αλλιώς τι, πώς θα εξελισσόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε ο Σινκλέρ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάποιον να δει κάποιον όταν εκείνος είναι αποφασισμένος να μην δει αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γερμανικά έχεις. Αγγλικά. Α, τίποτε τώρα. Γαλλικά. Πες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Kinu HDP, no my sa stále tvárime, že neexistuje. Namiesto uznania tohto prínosu jednoznačne... Jedno... Τώρα επανήλθε. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και πάλι διέκοψε η διακόπη διερμηνία. Λυπούμαστε πολύ. Στην αγροτικές κοινωνίες αυτό είναι κάτι που μπορεί πράγματι να εκτιμηθεί. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μαρινέσκου. Ο κύριος Ρόντιν, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε χώρα μπορεί βεβαίως να ορίζει το δικό της το ενεργειακό μείγμα. Αυτό όμως που κυρίως ενδιαφέρει είναι τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ε, ε, να μπορούμε να τις κλείσουμε όταν αποφασίζουμε κάτι τέτοιο. Όμως στη Λιθουανία και σε άλλες χώρες έχουμε πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν είναι πλέον ασφαλείς και οι οποίες ε, πρέπει να κλείσουν. Το πρόβλημα όμως είναι ο προγραμματισμός. Προγραμματισμός δεν υπάρχει. Κατόπιν τούτου λοιπόν ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, μέχρι το έτος 2013 να εκταμιεύσουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να πάψουν να λειτουργούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Ο προγραμματισμός όμως όπως σας είπα είναι ανεπαρκής και η Κομισιόν οφείλει να καταθέσει ανάλυση της αποδοτικότητας αυτών των μέτρων. Γιατί ε, θα πρέπει τα κράτη να μπορούν να αποδείξουν ότι πράγματι χρησιμοποίησαν τα κονδύλια όπως ακριβώς έπρεπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για τη χρηματοδότηση της προοδευτικής κατάργησης των πυρηνικών εγκαταστάσεων μας δείχνει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ με μια από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης ότι αυτή η προοδευτική κατάργηση αυτών των εγκαταστάσεων θα απαιτήσει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών κονδυλίων ακόμα και μετά το 2013. Δεν θα είναι δυνατόν για τις ενδιαφερόμενες χώρες να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους αυτή την προσπάθεια. Η Σλοβακία κάτω από την πολιτική πίεση Ευρωπαϊκής Ένωσης διέκοψε τη λειτουργία δύο, δύο μονάδων του πυρηνικού σταθμού της και σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ανάργειας στηρίθηκαν όλα τα κριτήρια ασφαλείας. Οι οικονομικές συνέπειες τέτοιων αποφάσεων είναι σημαντικά και συνεπάγονται τεράστιο κόστος για την προοδευτική αυτή κατάργηση των εγκαταστάσεων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτό το κόστος στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών 2013-2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν ώψη των πρόσφατων γεγονότων στην Ιαπωνία, η ενεργειακή πολιτική και η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα πολύ καυτό επίκαιρο θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καταστροφή στη Φουκοσίμα έδειξε πόση πολλή δουλειά θα χρειαστεί να γίνει για να δημιουργήσουμε ένα φιλικό προς το περιβάλλον και ασφαλές ενεργειακό δίκτυο. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ισία, αλλά για όλες τις υπήρους. Αν ε, ενεργειακές εγκαταστάσεις χρειαστεί να κλείσουν για λόγους ασφαλείας, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ασφαλείς πηγές ενέργειας. Ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα η προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το θέμα, που το παρουσίασε ο κύριο Αμαρουνέσκου, δεν μπορούμε εμεί να το συμμεριστούμε και να το εγκρίνουμε, διότι ε, χαρακτηρίζεται και υπάρχουν ακόμα αισθητέ επιπτώσει από τη Φουκοσίμα. Η προσέγγιση του θέματο από πλευρά συγητή είναι ισορροπημένη. Ε, εγώ βέβαια θέλησα να τον στηρίξω και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσον αφορά τη Λιθουανία, την Σλοβακία και τη Βουλγαρία, εκεί πρέπει να υπάρχει υπάρχει συνεπής αντιμετώπιση. μεταξύ όμως ε, θα πρέπει να αναλυφθούν και άλλες ε, δραστηριότητες όταν αποκαλούμε ε, δοκιμές αντοχής έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, δεν μπορεί να γίνει λάθος για λόγους που τους γνωρίζουμε όλοι μας. Τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν ήδη προβλεφτεί εδώ και καιρό, έχουν διασφαλιστεί. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα θα υπάρχει αίσιο τέλος και έτσι λοιπόν το όλο εγχείρημα θα έχει την κατάληξη που όλοι επιθυμούμε. Κύριος Μπαρτελότσι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των ε, επαρκών κονδυλίων για να διασφαλίσουμε τις ε, δραστηριότητες κλεισίματος των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι ένα θέμα το οποίο ήδη αντιμετωπίζεται από την νομοθεσία, το νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο. Βεβαίως υπάρχουν τα τελευταία γεγονότα που μας επηρεάζουν και όπως και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων που λήφθησαν υπόψη. Η έκθεση Μαρινέσκου ε, τη στηρίξαμε την έκθεση αυτή έχοντας κατά και ειδικέ περιπτώσεις ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία όταν προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και γι' αυτό το λόγο έτυχαν και ειδική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από συγκεκριμένε περιπτώσεις, το επιχείρημα αυτό ε, πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστικό έλεγχο των πυρηνικών αντιδραστήρων που υπάρχουν στην ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, είναι υψηλός ο των πυρηνικών αντιδραστήρων που πρέπει να προχωρήσουν στο αμέσως ε, στο εγγύ μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε μηχανισμούς ε, χορήγησης εγγύησεων και ε, κυρίως να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν. Είτε είναι ανάγκες προβλέψιμες είτε έκτακτες. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ στήριξα αυτό το θέμα ως επεπισμένος ε, αντίπαλος των πυρηνικών αντιδραστήρων όχι γιατί πιστεύω ότι η πάυση λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων θα αποφέρει πλεονεκτήματα στο σύνολο της κοινωνίας αλλά κυρίως διότι επιθυμώ να μην υπάρχουν τέτοιου είδους άλλες καταστάσεις. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε ε, πρόβλημα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουμε για τις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις Πρέπει λοιπόν να χειριστούμε το θέμα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην βασιζόμαστε μόνο σε αναχρονιστικές απόψεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι όσον αφορά αυτή την ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο θεωρητική και όλα πάνε καλά μέχρι να γίνει κάτι συγκεκριμένο. Τότε λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτόκολλο που είναι πολύ παλιό, 50 ε, ετών ε, ήδη διάρκεια ζωής που δεν προβλέπει τις ε, σημερινές καταστάσεις. Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ούτε τις τρομοκρατικές επιθέσεις ούτε τις ε, θεομηνίες που έλαβαν χώρα και δυστυχώς όλο και περισσότερο οι καταστροφές αυτές, οι σεισμοί συγκεκριμένα ε, λαμβάνουν χώρα όλο και περισσότερο. Και διακόπτω εδώ γιατί δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου κύριε Πρόεδρο. Ο κύριος Μετσάρος για ένα λεπτό. Σλοβακία επηρεάζεται από την πρόταση αυτή. Στην, ε, ε, ε, σύμβαση προσχώρησης είχαμε αναλάβει τον παροπλισμό των πυρονικών εγκαταστάσεων από το 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε οικονομικές ενισχύσεις για αυτή την προσπάθεια υπάρχουν, ε, υπάρχουν λίγες περιπτώσεις εμπειρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιες διαδικασίες παροπλισμού πυρονικών εγκαταστάσεων. Μπορεί να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Βεβαίως θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής, επαρκής χρηματοδότηση για να είναι, δυνατή, να είναι δυνατός ο ασφαλής παροπλισμός αυτών των εγκαταστάσεων. Η σχετική εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν φτάσει στη λήξη της χρήσιμης περίοδου τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα ώστε να αξιοποιηθεί στο μέλλον αποτελεσματικά αυτή η εμπειρία που θα αποκτηθεί. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, υπερψήφισα την έκθεση Μαρινέσκου ακριβώς γιατί στην ε, νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη υπάρχει μια βαριά κληρονομιά εξαιρετικά επικίνδυνων πυρηνικών αντιδραστήρων όπω στη βουλγαρία στη ρουμανία στη σλοβακία. όλα αυτά τα χρόνια όμω ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια ευρώ των ευρωπαίων πολιτών προκειμένου να εξυγχρονιστούν και να επιτύχουν παράταση τη ζωή του. πρόκειται ουσιαστικά για επιδότηση του πυρηνικού λόμπι που αναλάμβαναν τι μετασκευέ. η φουκουσίμα μα έχει δείξει για άλλη μια φορά ότι οι αντιδραστήρε αυτοί πρέπει να κλείσουν. όμω τέτοιε οικονομικέ προβλέψει δεν έχουν υπολογιστεί στο κόστο λειτουργία των αντιδραστήρων και αυτό αποτελεί μια τεράστια και σκανδαλώδη σκανδαλώδη επιχορήγηση για έναν επικίνδυνο δαπανηρό και ρηπογόνο τρόπο παραγωγής ενέργειας. και τώρα όμως αρκεί να αλλάξουμε πολιτική βούληση. μετατρέψτε άμεσα τις επιδοτήσεις για μετασκευές τους μη ασφαλείς αντιδραστήρες σε χρηματοδότηση για το κλείσιμό τους παγώστε όλους τους νέους αντιδραστήρες που σχεδιάζονται μεταφέρετε πόρους από τις χρηματοδοτήσεις της euratom και τι πλουσιοπάροχε επιχορηγήσει twitter εκτρέψτε τους πόρους που προορίζονται για μελέτες και κατασκευές νέων αντιδραστήρων σε μια οικονομία βασισμένη κατά 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το. 2050. είμαστε σε κατάσταση ανάγκης και πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθούμε. ευχαριστώ. Thank Sveikinu pranešėją Χαιρετίζω την έκθεση αυτή και συγχαίρω τον, τον εισηγητή για την έκθεση του. Η Λιθουανία μαζί με τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της με βάση τη συνθήκη προσχώρησης και παρόπλησε τους ε, αντιδραστήρες της. Εφαρμόστηκαν όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ελπίζουμε να προσάγουμε στη δικαιοσύνη εκείνους οι οποίοι δεν είχαν ε, εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις τους και θέλουμε να διαπραγματευτούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε ό,τι αφορά την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Συμφωνώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια με τον πιο διαφανή τρόπο, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο εξής. η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών στα σύνορα με τη, τη Λευκορωσία. Τελειώσαμε την έκθεση Μαρινέσκου και περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Μπάρμπαρα Ματέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ε, δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω ε, επεξήγηση ψήφου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να πω ότι το ε, φιλελεύθερο κόμμα στη Δανία είναι κατά του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Όμω, εφόσον έχει εγκριθεί και όταν θα υποβληθούν αιτήσει από τα διάφορα κρατημέλη και εφόσον πληρούνται οι προποθέσει για την απόκτηση αυτών των κονδυλίων, προφανώ θα πρέπει κανεί να το δεχτεί και να το υπερψηφίσει και γι' αυτό υπερψηφίσαμε. Κυρία Σίνκλερ, παρακαλώ. Thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα και αυτή την έκθεση, την έκθεση Ματέρα, αλλά και την έκθεση που είχε να κάνει με την Πολωνία, όχι γιατί τα έχουμε τις δύο αυτές χώρες, αντιθέτως, αλλά γιατί θα ήθελα να σας θυμίσω θέλω να σας πω ότι μου θυμίζουν τη δική μου περιφέρεια, στα West Midlands. Όμως εμείς συμβάλλουμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να σας μιλήσω για τα West Midlands. Να σας μιλήσω λίγο για αυτά. Έχουμε υψηλή ποσοστά ανεργίας. Η βιομηχανία μας αποδεκατίστηκε εν μέρη λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσχώρησης όλων αυτών των χωρών και της δημιουργίας εργοστασίων εκεί. Και μάλιστα το 2004 το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά δέχτηκε τεράστιο πλήγμα με τη διεύρυνση. Και τώρα έχουμε και μεγάλο κόστος ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες. Ε, μια άλλη δαπάνη που χρειάστηκε να αναλάβουν οι ψηφοφόροι μου είναι η εξή. Εμείς συμβάλλουμε στα, ε, στη φροντίδα των παιδιών εργαζομένων που έρχονται από τις, ανατολικ... τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Μιλάμε για 48 εκατομμύρια στερλίνες και μάλιστα ημερησίως, οι οποίες καταβάλλονται. Ευχαριστώ. Mr. Kelly. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ στήριξα τις εκθέσεις αυτές και θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στους εργαζόμενους στη Δημοκρατία της Τσεχίας και στη Πολωνία. Και με πολύ μεγάλη λύπη ακούω τους προλαλήσαντες και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τι συνέβη στη δική μου περιφέρεια με την Waterford Crystal. Θα πρότεινα λοιπόν το κράτος μέλος να είναι σε θέση να υποβάλει προτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των κονδυλίων και την καλύτερη βοήθεια προς τους εργαζομένους. η ανεργία είναι ένα πρόβλημα και πιστεύω ότι μπορεί να καταπολεμηθεί με αυτόν τον τρόπο και να βελτιωθεί και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, καλώς. Πάμε στην έκθεση Σβένσον, ο κύριος Ρέντερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η βία κατά των γυναικών, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο και βεβαίως ε, πρέπει να τοποθετηθούμε επί του θέματος αυτού και ως άνθρωποι και ως πολιτικοί. Οφείλουμε να λάβουμε θέση για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα η Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην παρουσίαζε έναν ατελείωτο κατάλογο ετοιμάτων. Εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες πρωτοβουλίε, αλλά καλύτερα να συζητάμε στοχευμένα και να λέμε ποιες πρωτοβουλίε μπορούν να αναλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λείπει είναι, όπως σας είπα, η στόχευση. Και αν είχαμε προτεραιότητες, τότε θα ήμασταν και πιο αποτελεσματικοί. Και αυτό θεωρώ ότι θα βοηθούσε και τις γυναίκες και θα προσέφερε και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις πρωτοβουλίες που προτείνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η βία κατά των γυναικών ε, δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα. Πρόκειται για έγκλημα που πρέπει να διωχθεί πρέπει να θέσουμε τέρμα στη σιωπή. Σε ό,τι ο σεβασμός της πολιτισμού και της θρησκείας είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να είναι ε, αφορμή για εμπορία, ενδοοικογενειακή βία, υποχρεωτικούς γάμους, ε, ε, γενετικούς ε, ε, ακροτηριασμούς των γενετικών οργάνων, των γενετικών οργάνων των γυναικών κλπ. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ε, με όλα τα πολιτικά κόμματα για να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Υποστηρίζω την αρχή και τα περισσότερα στοιχεία της πρότασης. Αλλά μέτρα ποινικά και δικαστικά θα πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό κάνουμε στη Σουηδία. Η βία ε, είναι ένα από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται το κόμμα μου ώστε να συνδυτοποιήσει το κοινό και να δώσει υπευθυνότητα στις γυναίκες και να εξασφαλίσει το σεβασμό ε, όλης της κοινωνίας για αυτό το φύλλο. Η κυρία Κώστα Σίλβια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπερψηφίζοντας αυτήν την έκθεση του κυρίου Σβένσον, όπως πολύ σωστά ελέγχθη και από άλλους συναδέλφους, της κυρίας Σβέντσον, με συγχωρείτε, ε, ζητάμε πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσα στο 2011 να ε, προβεί σε μια ανακοίνωση στρατηγικής στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών. Να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να περιλαμβάνει όλα τα είδη βίας ε, της σεξουαλικής, της κατοίκων βίας, ε, τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Πιστεύω ότι αυτές οι νέες μορφές της βίας είναι εκείνες που οδηγούν στο να βγαίνει στον τύπο όλη αυτή η βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών και αυτό αυτό είναι και μία απειλή για τις γυναίκες ε, ε, στον χώρο εργασίας. Έτσι λοιπόν υπάρχει και η οδηγία για την παράνομη διακίνηση ανθρώπινων όντων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και μία άλλη οδηγία εφόσον έχει εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και το πρόγραμμα της Στοχάλμης να εκδώσουμε μία συγκεκριμένη οδηγία για το θέμα αυτό. Κύριε Ρονσούλη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μέχρι αυτές οι μορφές βίας κατά των γυναικών να εξαλειφθούν, δεν θα μπορούμε ποτέ να πούμε ότι θα έχουμε μια σύγχρονη και δημοκρατική κοινωνία. Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφει την προσοχή του σε αυτό το βίαιο φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς παραμένει και τραγικά επίκαιρο. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, μία στις πέντε γυναίκες δέχεται σεξουαλική ή σωματική βία κατά διάρκεια της ζωής της. Μάλιστα για τις γυναίκες από 15 μέχρι 44 ετών η βία είναι ο πρώτος, ε, πρώτο αίτιο που οδηγεί στο θάνατο, περισσότερο από τον καρκίνο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια μόνιμη δραστηριοποίηση που θα οδηγήσει στο να συσταθεί ένα παγκόσμιο νομικό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν όλες οι μορφές βίας που ασκούνται κατά των γυναικών. Σήμερα πρέπει να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα, γιατί ο στόχος ε, είναι ένας, ότι δεν θα πρέπει πλέον να ασκούνται τέτοιες μορφές βίας εις βάρος των γυναικών. Η κυρία Μπιλμπαμπαράντικα. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Η βία κατά των γυναικών είναι άμεση απόρρια της διάκρισης. Εξού και μας χρειάζεται μια ενιαία ολοκληρωμένη πολιτική που να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά των κακοποιημένων γυναικών. Θα πρέπει να έχουν δωρεάν νομική και ιατρική περίθαλψη, θα πρέπει να έχουμε κέντρα που να διευκολύνουν την αυτονομία τους, ε, ειδικά πρωτόκολλα ενημέρωσης, ειδική ενημέρωση του, των αστυνομικών αρχών αλλά και των υγειονομικών αρχών. Και χρειαζόμαστε και συλλογή στοιχείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα και να εφαρμόσουμε σωστότερα τις πολιτικές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βανχέκε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας για την έκθεση Σβένσεν δεν έλαβα μέρος στην ψηφοφορία Βεβαίω ε, είναι απαράδεκτη βία κατά των γυναικών. Απέσχα από την τελική ψηφοφορία ωστόσο επειδή πιστεύω ότι αυτή η έκθεση παραβιάζει κατ' επανάληψη την αρχή της επικουρικότητας την οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία και δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το επιθυμητό. Επίσης δεν δέχομαι την ε, το, οδηγίες για το ποια είναι η πολιτική, πολιτικά ορθή συμπεριφορά. Αναφέρεται το Ισλάμ κατά επανάληψη. Μιλάμε για μια θρησκεία με πεπαλωμένες ιδέες η οποία οπωσδήποτε παίζει σημαντικό ρόλο στις πράξεις βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι κάτι το πάρα πολύ φυσικό για το Ισλάμ η κυρία Ζαμπόρσκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έκθεση Σβένσον συμβάλλει ιδιαίτερως ε, στη συζήτησή μας. Φυσικά και κατακρίνουμε τη βία και κυρίως ενάντια των εγκύων γυναικών. Πιστεύω ότι κάνουμε ένα βήμα προς τα πέρα, προς, τα εμπρός. Έχω προσπαθήσει πολύ ε, να συμβάλλω στην ε, ε, στην προστασία των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Ωστόσο, η έκθεση δεν μας βοηθάει απολύτως να ε, ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Θεωρώ ότι η άμβλωση είναι βία που ασκείται εναντίον των αγέννητων παιδιών. Και όταν ε, ε, ε, χαράσουμε τη στρατηγική μας ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει περισσότερο ώστε να επιτευχθεί ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και των δικαιωμάτων των αγέννητων παιδιών. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίνκλερ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της έκθεσης Svensson προφανώς καταδικάζω τη βία κυρίως τη βία κατά των γυναικών. Γιατί λοιπόν ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης. Ψήφισα κατά επειδή όπως είπε ένα συνάδελφος πριν από λίγο μας φέρνει, οδηγεί πίσω στα θέματα της πολιτικής ευπρέπειας και στη δεκαετία του 1970. Δεν ξέρω αν θέλουμε να επανέλθουμε στη δεκαετία του 1970. Και με προβληματίζει το το, το, θέμα της εγκληματικής πράξης, το στοιχείο της εγκληματικής πράξης που θέλουν να προωθήσουν διότι μιλάμε για την άσκηση ποινική δίωξης και την οποία εκτείνουμε σε όλο και περισσότερους τομείς. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή η επιλογή αυτής της έκθεσης παρόλο που πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ουσιαστικές ενέργειες και παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσεις ψήφου, λύεται η συνεδρίαση, θα επανεληφθεί στις 3 το απόγευμα.